το καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να, προ... να μας ε, υποβάλει ένα αριθμιστικό πλαίσιο. Ένας μεγάλος αριθμός στοιχείων είναι απαραίτητος για τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και Έχουμε σαφώς την Cambridge Analytica και την ε, Clearview που είναι προφανή παραδείγματα για την ε, χρήση και κατάχρηση δεδομένων. Ε, η χειραγώγηση δεδομένων είναι σοβαρή απειλή για τις δημοκρατίες μας. Η ψηφιακή επανάσταση δεν είναι τίποτα νέο και είναι υπό εξέλιξη εδώ και χρόνια. Όμως διαρκώς πρέπει να μπορούμε να βρούμε νέες απαντήσεις στις νέες τεχνολογίες. Και να θυμίσω επίσης ότι ο κανονισμός GDPR, συνάδελφοι για παράδειγμα, μας πήρε σχεδόν έξι χρόνια μέχρι ότου εγκριθεί. Και αυτό μας δείχνει πως η τεχνητή νοημοσύνη, η εποπτεία και η αναγνώριση προσώπου ήδη χρησιμοποιούνται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να βιαστούμε για να τα δομήσουμε σωστά. Είναι καθήκον μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκπρόσωποι των λαών του Ευρωπαϊκού της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα μείνει κανείς πίσω. Η Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Ατζέντα θα πρέπει να βασίζεται στις ευρωπαϊκές μας αξίες και να προσφέρει ευκαιρίες για όλους. Ευχαριστώ. Thank you very much. And now I would like... Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος στο Συμβούλιο. Ε, Υφυπουργός ε, κυρία Μπρινιάτσκ. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να συμμετάσχω σε αυτή τη συζήτηση. Είναι σημαντικό να προβληματιστούμε για το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διασφαλίσει ότι μια διαρκώς όλο και πιο ψηφιοποιημένη Ευρώπη μπορεί ε, να είναι και κοινωνική. Η, κοινωνία κοινωνική οικονομία της αγοράς είναι πλεονέκτημά μας, ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα, αλλά θα πρέπει να την προετοιμάσουμε, να την προσαρμόσουμε στον μεταβαλλόμενο κόσμο. Η ψηφιοποίηση είναι μια οριζόντια διαδικασία που παρουσιάζει και ευκαιρίες και κινδύνους μπορεί να οδηγήσει σε δημιουργία νέων ποιοτικών θέσεων εργασία, μπορεί να αυξήσει την αποδοτικότητα, να βελτιώσει την ευημερία των εργαζομένων και με αυτόν τον τρόπο ε, να βοηθήσει τη συμφιλίωση επαγγελματική και προσωπική ζωή. Επίση, μπορεί να προσφέρει καινούριε ευκαιρίε σε ανθρώπου ε, από ευάλωτε ομάδε και ανθρώπου με αναπηρίε. Όμω, όπω και όλε οι αλλαγέ, έχει και, ενέχει και κινδύνου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, πρωτοστατεί στο να διασφαλίσει ότι αυτές οι αλλαγές θα οδηγήσουν και σε κοινωνικές βελτιώσεις και ενώ θα προστατεύσει ταυτόχρονα και αυτούς που τείνουν να μείνουν πίσω ή να εξαιρεθούν. Ε, από το 2019 έχουμε την ανακοίνωση για το μέλλον της ε, Ευρώπης, την οποία υποστηρίζουμε. Σήμερα όμως έχουμε και τρεις πτυχές που έχουν σχέση με την ψηφιοποίηση και τις και οι οποίε ε, είναι σίγουρο ότι θα επηρεάσουν πολύ τη ζωή μα. Πρώτον, τα προσόντα. Δεύτερον, η οικονομία των πλατφορμών. Τρίτον, οι κοινωνικέ επιπτώσει της ψηφιοποίηση. Σε ό,τι αφορά τα προσόντα, ε, τα, η ψηφιοποίηση επηρεάζει με δύο τρόπου. Πρώτον, αυξάνει την ζήτηση ε, για εργαζόμενους με συγκεκριμένα και αυξημένα προσόντα. Δεύτερον, μερικές, μερικά επαγγελματα θα αλλάξουν ή θα εξαφανιστούν. Ε, ο κίνδυνος είναι η δημιουργία μεγαλύτερης ανεργίας και ανισοτήτων. Ε, πολύ συχνά θα χαθούν οι ενδιάμεσες θέσεις εργασίας. Ε, πολύ συχνά επίσης τα σημερινά προσόντα δεν θα ταυτίζονται με τα προσόντα που οποία θα απαιτούνται σύντομα στο μέλλον. Ειδικεύση σε τεχνολογία, μαθηματικά, επιστήμες κλπ. Επίσης είναι πιθανό να επιδεινωθεί το πρόβλημα ε, της ανισότητας μεταξύ των δύο φύλων. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη λοιπόν το πώς ε, η ψηφιακή επανάσταση επηρεάζει τη ζωή του ανθρώπου από την παιδική του ηλικία. Κανείς δεν πρέπει να μείνει εκτός. Και οι άντρε και οι γυναίκες χρειάζονται για να καλυφθούν οι ελλείψεις στα προσόντα σχετικά με την κοινωνία της πληροφορίας. Ε, το εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να καταπολεμήσει τα ταμπού ε, και τις προκαταλήψεις, ε, τα στερεότυπα. Θα πρέπει επίση να προσαρμοστεί το εκπαιδευτικό σύστημα στι ανάγκε του μέλλοντο και οι κοινωνικοί εταιρείε έχουν να παίξουν σημαντικό ρόλο. Να βοηθήσουν έτσι ώστε να διατηρηθεί η προσαρμοστικότητα τη της ε, εργασιακή δύναμη. το δεύτερο, οι πλατφόρμες φέρνουν πολύ κοντύτερα και σε άμεση επαφή τους προμηθευτές με τους πελάτες. Πολλές ε, πλατφόρμες ε, θα απασχολούν έμεσα ανθρώπους ε, οι οποίοι θα εξαρτώνται από τη λειτουργία της πλατφόρμας. Εκεί έχουμε θέματα αμοιβή, κοινωνικής προστασίας, δικαιωμάτων σε άδεια κλπ. Ο αποτελεσματικός κοινωνικός διάλογος σε όλα τα επίπεδα είναι απόλυτος απαραίτητος για να διασφαλίσουμε ότι το μέλλον θα είναι δίκαιο και ισότιμο. Είναι δύσκολο όμως οι εργαζόμενες πλατφόρμες να, ε, να δημιουργήσουν συνδικάτα ή όργανα που τους εκπροσωπεί γιατί δεν γνωρίζονται και δεν εργάζονται μαζί στον ίδιο χώρο. Αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ίδιε συνθήκε εργασία για όλου, ανεξάρτητα από αλλαγέ στα σχήματα ε, πρόσληψης ε, και απασχόληση. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, ήδη έχει γίνει ένα πρώτο βήμα με την οδηγία για τις ε, διαφανείς και προβλέψιμες συνθήκες εργασίας. Η σύσταση για την ε, κοινωνική προστασία αυτοπασχολούμενων που υιοθετήθηκε το Δεκέμβριο από το Συμβούλιο αναφέρεται ρητά στους εργαζόμενους σε πλατφόρμες και συστήνει στα κράτη-μέλη να προσφέρουν κοινωνική προστασία σε όλους ακόμα και τους αυτοπασχολούμενους. Επίσης το Συμβούλιο υπογράμμισε ότι οι πολιτικές κοινωνικές προστασίας θα πρέπει ε, να ακολουθούνται και από αντίστοιχε πολιτικές ε, μισθολογικές πολιτικές έτσι ώστε και αυτοί που ε, ακολουθούν και τα καινούργια μοντέλα εργασίας να μπορούν να αποφεληθούν από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Επίσης το Συμβούλιο έχει αναφέρει ότι αυτοί οι εργαζόμενοι στις καινούργιες θέσεις εργασίας θα πρέπει να προστατεύονται σε ό,τι αφορά την υγεία και την ασφάλεια τους. Ανεξαρτήτως ε, τη, της μορφής εργασιακής σχέσης. Επίσης έχει υπογραμμίσει το Συμβούλιο ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί αποτελεσματικά η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, ακόμα και για τι νέε μορφέ εργασία. Θα πρέπει να καταλάβουμε καλύτερα το πώ λειτουργούν οι πλατφόρμε, έτσι ώστε να επεξεργαστούμε καινούριε πολιτικέ. Από αυτή την έννοια περιμένουμε ε, την, ε, την Σύνοδο Κορυφή ε, για του εργαζόμενου πλατφόρμες που θα διοργανώσει η Γερμανική Προεδρία τον Οκτώβριο του τρέχοντο έτου. Τρίτον, την κοινωνική επίδραση των πλατφορμών τη ψηφιοποίηση. Οι αλλαγέ λόγω τη ψηφοποίηση έχουν διάφορε επιπτώσει. Αφενό, οι εργαζόμενοι μπορούν να, είναι πιο ελαστικ... να, να εργάζονται πιο ελαστικά. Απ' την άλλη μεριά, ε, πολύ συχνά είναι αναγκασμένοι, είναι συνεχώς ε, συνδεδεμένοι με την εργασία τους. Ε, το ίδιο μπορεί να συμβεί, παρόμοιες ε, θετικές και αρνητικές συνέπειες μπορούμε να δούμε και στους ανθρώπους με αναπηρίες. οι εργοδότες έχουν καλύτερα εργαλεία για να παρακολουθούν την αποδοτικότητα επίσης. Η τεχνολογική εξέλιξη είναι αναπόφευκτη. Θα πρέπει να την αγκαλιάσουμε. Ε, χρειάζεται να υιοθετήσουμε καιρούς τεχνολογίες. Αυτό θα μας δώσει περισσότερο έλεγχο για το προς τα που κινούμαστε, κινούμαστε αλλά θα πρέπει να κινηθούμε με βάση τον άνθρωπο θα πρέπει οι αποφάσει μα να είναι τεκμηριωμένε, χωρί να ξεχνάμε ότι η κοινωνική οικονομία τη αγορά είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα τη Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον Επίτροπο Σμιτ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, η ψηφιακή ε, μεταρρύθμιση θα έχει και θα έχει ήδη αντίκτυπο άνευ προηγουμένως στις οικονομίες μας, στις κοινωνίες μας, τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε, επικοινωνούμε ή καταναλώνουμε. Το θέμα της απασχόλησης είναι βέβαια στο επίκεντρο των προβληματισμών. Πόσες θέσεις απασχόλησης θα χαθούν και θα αντικατασταθούν εκεί οι άνθρωποι από ρομπότ. Αυτό που είναι ήδη βέβαιο είναι ότι οι περισσότερες θέσεις απασχόλησης θα αλλάξουν νέες, νέου είδους δουλειές θα εμφανιστούν, ενώ άλλες θα εξαφανιστούν και άλλες ε, θα αλλάξουν ε, ρηξικέλευθα. Η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική θα δημιουργήσουν μόνες τους γύρω στα 60 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης στον κόσμο στη διάρκεια των επόμενων 5 ετών υπολογίζεται. Και ήδη σήμερα, γι' αυτό αναφέρθηκε ήδη, γύρω στο 1 εκατομμύριο θέσεων στην πληροφορική είναι κενές γιατί δεν υπάρχουν αρκετοί υποψήφια με τις απαραίτητες γνώσεις. Είναι πολύ σημαντικό γι' αυτό πολλές εταιρείες, κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν βρίσκουν ε, ε, το κατάλληλο προσωπικό με τα απαραίτητα προσόντα. Και αυτό είναι μεγάλη πρόκληση για τις πολιτικές απασχόλησης και εκπαίδευσης. Κυρίες ε, και κύριοι, κυρία Πρόεδρε, δράσαμε με το να ιδρύσουμε το Ταμείο Δίκαιη μετάβαση όσον αφορά την πράσινη μετάβαση για τις περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε ενισχύοντας τις κοινωνικές πολιτικές και τις πολιτικές απασχόλησης για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τις άλλαγέ που αναμένουμε από την ψηφιοποίηση. Υπάρχουν και έχει ήδη αναφερθεί πολλές καλές ευκαιρίες, αλλά υπάρχουν και κίνδυνοι του να αυξηθούν οι ανισότητες ε, και η επισφάλεια. Πάνω από το 90% των θέσεων εργασίας αυτή τη στιγμή απαιτούν κάποιο επίπεδο ψηφιακών δεξιότητων, όπως και η συμμετοχή στην κοινωνία γενικώ. Όμως, 43% του πληθυσμού έχουν ανεπαρκές επίπεδο ψηφιακών δεξιότητων. 17% δεν έχουν καθόλου. Τον επόμενο μήνα θα προτείνουμε ένα νέο πρόγραμμα για τις δεξιότητες για να αντιμετωπίσουμε ακριβώς αυτό το θέμα με συγκεκριμένα μέσα. Και η πρόκληση είναι τεράστια, γιατί σύμφωνα με πολλές προβλέψεις οι μισοί Ευρωπαίοι εργαζόμενοι, πάνω από 120 εκατομμύρια άνθρωποι, θα πρέπει να αλλάξουν ή να αυξήσουν τις δεξιότητες τους. Έχουμε λοιπόν τρεις κύριους στόχους. Ο πρώτος είναι να έρθουμε σε επαφή με τους εργοδότες για να εκπαιδεύσουν περισσότερο τους εργαζόμενους. Για το σκοπό αυτό θα συντάξουμε ένα σύμφωνο δεξιοτήτων που θα δεσμεύει τις επιχειρήσεις για να επενδύουν στους εργαζομένους τους. Δεύτερον, πρέπει να αυξηθούν οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερα. Και τρίτον, πρέπει να ενδυναμώσουμε τους ανθρώπους για να επενδύουν οι ίδιοι στα προσόντα τους και τις δεξιότητες τους. Πολλές από τις πρωτοβουλίες μετά το 2020 θα αφορούν ακριβώς τις προκλήσεις της ψηφιοποίησης. Το ταμείο αυτό θα στηρίζει έργα όπως η δημιουργία ηλεκτρονικών σχολείων με δασκάλου οι οποίοι θα εκπαιδεύουν ανέργου για δουλειέ στον τομέα της πληροφορική. και εργαζόμαστε σε μια ενισχυμένη εγγύηση για την νεολαία να υπάρξει μια πολύ σοβαρότερη κάλυψη των ψηφιακών δεξιοτήτων. Οι άτυπε μορφές εργασίας αυξάνονται και συνοδεύονται από ευελικτές και συχνά ανεπαρκείς συνθήκες ε, εργασίας ε, μειωμένη πρόσβαση στην κοινωνική προστασία, απουσία κοινωνικού διαλόγου και συλλογικών διαπραγματεύσεων. Αυτό αποτελεί πρόκληση για τα συστήματα εργατικού δικαίου και κοινωνικής προστασίας και απαιτεί να επανεξετάσουμε τα υφιστάμενα μοντέλα για να διασφαλίσουμε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, συμπερίληψη και υψηλό επίπεδο κοινωνικής προστασίας η ψηφιοποίηση αλλάζει το πώς βλέπουμε την δουλειά, τις σχέσεις εργαζομένων εργοδοτών και τον χώρο εργασίας. Και είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρξει σαφήνεια στον νέο κόσμο της εργασίας. Οι νέες τεχνολογίες επίσης καταργούν τη διάκριση μεταξύ ιδιωτικού βίου και εργασίας. Υπάρχουν έτσι νέοι κίνδυνοι για τη σωματική και ψυχική υγεία. Άρα το δικαίωμα να αποσυνδεθούμε είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε. Η χρήση των δεδομένων έχει οδηγήσει σε διαχείριση με βάση τους αλγόριθμους και αύξηση της διαχείρισης του προφίλ. Αυτά μπορούν να αυξήσουν την παραγωγικότητα αλλά και τον έλεγχο και την εποπτεία των ατόμων και των εργαζομένων γύρονται θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος σε αυτά στο πλαίσιο της ρύθμισης της τεχνητής νοημοσύνης. Χρειαζόμαστε ψηφιακές τεχνολογίες προσβάσιμες και διαλειτουργικές για να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες της ψηφιοποίησης για να αυξηθεί η αυτονομία των ατόμων με αναπηρία και να αυξηθεί η συμμετοχή τους στην κοινωνία και στην οικονομία. Ο ψηφιακό μετασχηματισμός πρέπει επίσης να αποτελέσει μια ευκαιρία στο πλαίσιο της δημογραφικής πρόκλησης που αντιμετωπίζουμε, ειδικά σε σχέση με την γύρανση του πληθυσμού και των περιοχών της υπαίθρου. Επίσης, πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στο χάσμα των φύλων που υπάρχει στον ψηφιακό κόσμο. Η Ευρώπη πρέπει να είναι ένας παίκτη ανταγωνιστικός και καινοτόμος. Οι νέες πρωτοβουλίες για τον ε, νόμο περί ψηφιακών υπηρεσιών θα παίξουν βασικό ρόλο μειώνοντας επίσης τον κίνδυνο διακρίσεων. Τον Σεπτέμβριο στις 23 του μηνός μαζί με την κυρία Βεστάγκερ θα οργανώσουμε μια σύνοδο κορυφής για την εργασία σε πλατφόρμες όπου θα συζητήσουμε το πώς ακριβώς θα βελτιωθούν οι συνθήκες εργασία στις διαδικτυακέ πλατφόρμες. Πέρα από αυτό, έχουμε ξεκινήσει την διαδικασία που σε ένα σχέδιο δράσης για έναν ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Επειδή οι αρχές του πυλώνα θα πρέπει επίσης να ισχύουν πλήρως και για τον νέο ψηφιακό κόσμο εργασίας. Ο πυλώνας αυτός θα πλαισιώνει την κοινωνική μας στρατηγική για να έχουμε μια μετάβαση σε μια κοινωνία ουδέτερη κλιματικά, η οποία θα είναι και κοινωνικά δίκαιη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Τώρα, εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων, για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ο κύριος Ράντικε για 1,5 λεπτό. Ναι. Κυρία Αντιπρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον κύριο που έθεσε το θέμα στην ημερήσια διάταξη. Την σύνδεση δηλαδή της ε, κοινωνικής διάστασης και της συζήτηση που κάνουμε εδώ για κοινωνική Ευρώπη με το σημαντικό αυτό θέμα της ψηφιοποίησης. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Συμφωνώ με αρκετά από αυτά τα οποία ήδη ακούστηκαν και στη συζήτηση που θα γίνει δεν πρέπει να ξεχνάμε το ότι τα τελευταία 20 χρόνια είχαμε τεράστιες αλλαγές στον κόσμο της εργασίας. Αφενός, οι σχέσεις εργασίας έχουν αλλάξει πλήρως. Έχουμε cried workers, glid workers, ε, εργασία η οποία είναι σε ετοιμότητα, αλλά έχουμε και τελείως διαφορετικούς τρόπους εργασίας. Έχουμε τις συσκευέ αυτές ε, στη τσέπη μας και ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να σχολάσουμε κάποια στιγμή να σταματήσουμε να δουλεύουμε όταν έχουμε συνέχεια μαζί μας το τηλέφωνο. Γι' αυτό λοιπόν στη συζήτηση αυτή που κάνουμε σημαντικό είναι να δούμε ήρεμα και να αξιολογήσουμε ευκαιρίες και κινδύνους, να δούμε πού πρέπει να παρεύουμε, πού πρέπει να στηρίξουμε. Γιατί για μένα είναι σαφές, είτε μιλάμε για τεχνολογία, είτε για οικονομία, όλα αυτά υπηρετούν τον άνθρωπο. Αυτό πρέπει να είναι η εποδός του πολιτικού μας έργου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, η κυρία Γιονγκέριους. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. σε 10 χρόνια θα έχει αλλάξει τελείω ο κόσμος της εργασίας χάρη σε τεχνολογίες οποίες ακόμα δεν γνωρίζουμε. Βεβαίω ε, θα πρέπει αυτά να πάνε προ σωστή κατεύθυνση. Τώρα έχουμε νέες κατηγορίες εργαζομένων σε πλατφόρμα όπως οι εργαζόμενοι του Uber στο Άμστερνταμ που ζητάνε παραδείγματος χάρη νορμάλ ώρες εργασίας, αλλά και να μπορούν να επηρεάσουν τις βαθμολογίες που τους βάζουν οι πελάτες, γιατί μια κακή βαθμολογία τους καταστρέφει και θα πρέπει να μπορούν να αποφασίζουν και το ρυθμό της εργασίας τους. Μπορούν λοιπόν να γίνουν τα πράγματα διαφορετικά. Η ψηφιοποίηση θα πρέπει να περιστρέφεται γύρω από τον άνθρωπο με αξιοπρεπές εισόδημα και καλή δουλειά. Θέλουμε λοιπόν να συζητήσουμε για τους κανόνες, ε, για τους εργαζόμενους στις ε, πλατφόρμες και αναμένουμε την συνάντηση στις 22 Σεπτεμβρίου. Thank you very much. Ευχαριστώ. Εκ μέρους του Renew Europe, ο κ. Πισλάρου. Για δύο λεπτά. Πρόεδρε, κύριε Επιτροπέ, συνάδελφοι. Εμείς οι Ευρωπαίοι πιστεύουμε στις δημοκρατικές αρχές. Και μια δημοκρατία που βασίζεται στους πολίτες της σημαίνει ότι είναι μια κοινωνική δημοκρατία. Και πρέπει να βοηθήσουμε τους πολίτες μας να υποφεληθούν από τις ευκαιρίες που δίνονται. Τους το οφείλουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι γνωστή ως πρωταθλήτρια στην νομοθεσία και τους κανονισμούς, τις οδηγίες κλπ. Όμως ο νόμος, η νομοθεσία δεν είναι αρκετή πια πρέπει να δράσουμε έτσι ώστε να μετασχηματιστεί η Ευρώπη και σε ένα πρωταθλητή της καινοτομία. Δυστυχώς υστερούμε. Πώς θα γίνει όταν ένας από τους... Ε, ένας, ε, το 20% των Ευρωπαίων πολιτών μας ε, δεν έχουν τα κατάλληλα προσόντα. Τα προσόντα είναι πάρα πολύ σημαντικά έτσι ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν σε μια αγορά εργασία που μεταβάλλεται και η ίδια είναι πολύ ρευστή. Αυτή είναι η προτεραιότητα, η κύρια προτεραιότητα για το αύριο. Θα πρέπει να απαντήσουμε στι καθημερινές ανησυχίες των πολιτών μας, δίνοντας την ευκαιρία να προσαρμοστούν στις προκλήσεις και να επωφεληθούν των ευκαιριών. Πώς? Το καλύτερο είναι επενδύοντας στους ίδιους ανθρώπους. Χρειαζόμαστε επενδύσεις που ε, θα συνδυάζουν ε, συνεισφορά του δημόσιου τομέα και του ιδιωτικού τομέα με τρόπο ώστε να βοηθήσουμε τους πολίτες μας να ξεπεράσουν τις ανισότητες που ενδεχομένως θα δημιουργήσει η τεχνολογική εξέλιξη. Χρειάζεται ε, ένα σχέδιο συνεργασίας δημο, ε, κρατικού και ιδιωτικού, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ε, έτσι ώστε να προωθήσουμε την ψηφιακή εκπαίδευση. Τι περιμένουμε. Θα ήθελα λοιπόν να επενδύσουμε στην ψηφιακή εκπαίδευση, για μια πιο κοινωνική και η Ευρώπη και να διευρύνουμε τις ευκαιρίες που δίνει η ψηφιακή οικονομία έτσι ώστε τα παιδιά, τα παιδιά του αύριο να μπορέσουν να επωφεληθούν πλήρως. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, εκ μέρους του, ε, της ομάδας της ε, Ταυτότητας και Δημοκρατίας, κυρία Ζαμέ. Πρόεδρε, μια κοινωνική Ευρώπη σε ένα ψηφιακό κόσμο είναι εντυπωσιακό το ότι Κανείς δεν μιλάει απλώς για την κοινωνική Ευρώπη. Πριν προχωρήσουμε στον ψηφιακό κόσμο, υπάρχει αυτή η, ψηφιακή Ευρώπη, η κοινωνική Ευρώπη. Η Επιτροπή ΕΜΠΛ το γνωρίζει πολύ καλά ότι ο συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, για παράδειγμα, είναι πολύ δυσχερή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, πολλοί πιστεύουν ότι θα ήταν πανάκια η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά η τεχνητή νομοσύνη και η ρομποτική παρουσιάζουν και πολλούς κινδύνους. Σίγουρα δεν είναι πανάκια. Υπάρχουν πάρα πολλά project τα οποία θα μπορούσαν να πλήξουν την εθνική κυριαρχία. Η προστασία των δεδομένων ε, είναι, δεν, δεν είναι εξασφαλισμένη καθόλου. Το αντίθετο σε σχέση με την Κίνα και τις ΗΠΑ. Η συλλογή δεδομένων κοινωνικής ασφάλισης, ε, αν πέσει σε, σε λάθος ε, χέρια, μπορεί να δημιουργήσει σοβαρότατα προβλήματα. Να χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς κλπ. Προφανώ είμαστε υπέρ τη ε, συνεργασία μεταξύ των μελών, υπέρ τη ψηφιοποίηση κλπ. Αλλά αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε πιο επίγοντα πράγματα, όπως το κοινωνικό dumping, το φορολογικό dumping ή την παγκοσμιοποίηση που Θα πρέπει αυτά να ρυθμίσουμε πρώτα. Ευχαριστώ. Εκ μέρους των Πρασίνων, για ένα λεπτό, ο λόγος στην κυρία Γκίσε. Ähm, Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, το αναφέρατε μόλις. Οι ψηφιακές τεχνολογίες ε, παραμελούν τους ε, φτωχούς ε, και ειδικά αυτούς οι οποίοι εξαρτώνται από τη στήριξη της κοινωνίας. Την προηγούμενη εβδομάδα απαγορεύτηκε σε δικαστήριο ένα τέτοιο σύστημα. Το ΣΥΡΙ, το οποίο στην Ολλανδία ε, προσπαθούσε να προβλέψει με έναν μυστικό αλγόριθμο ποιοι ήταν πιθανότερο να κάνουν απάτες για τα επιδόματα. Αλλά το κοινωνικό κράτος λέγεται κοινωνικό γιατί ακριβώς βοηθάει τους ανθρώπους, όχι να τους κατασκοπεύει. Δεν έχει καμία δουλειά να κάνει κάτι τέτοιο. Αντίθετη ερώτηση. Γιατί δεν σκέφτηκε κανείς να δει πού ακριβώς ε, δίνει τα λεφτά το κράτος, ε, γιατί ακριβώς χρησιμοποιείται τεχνητή νοημοσύνη για φοροδιαφυγή. Αυτά τα πράγματα χρειαζόμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τους Ευρωπαίους ε, συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές η κυρία Ραφάλσκα για ένα λεπτό. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, διαρκώς ακούμε ότι ο άνθρωπος πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της ψηφιακής οικονομίας. Ωστόσο, όλες οι διάφορες προκλήσεις θα πρέπει να συνδυαστούν με την κοινωνική πρόνοια και πρέπει αυτές οι αλλαγές να είναι θετικές για τους, για τους ε, υπαλλήλους μας. Η ρομποτική και η τεχνητή νομοσύνη θα δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης, αλλά εκεί ενεργούνται κίνδυνοι. Θέλουμε αυτές οι νέες θέσεις να είναι υψηλής ποιότητας, θέλουμε νέες μορφές απασχόλησης και θέλουμε αυτού του είδους απασχόληση να είναι ελκυστική. Ωστόσο, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πως οι ευκαιρίες αυτές θα είναι ανοιχτές για όλα τα κρατημέλη και ότι δεν θα υπάρξει κοινωνικός απο... Ε, ε, ψηφιακός με αποκλεισμός, ειδικά όταν πρόκειται για τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ε, στηρίξει όλες τις περιφέρειες. Οι αλλαγές αυτές είναι αναπόφευκτες. Οι κανονισμοί δεν μπορούν να κάνουν ε, όλη τη δουλειά. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε κοινωνική ασφάλιση, καλές συνθήκες εργασίας και κοινωνική πρόνοια για τους εργαζόμενους μας. Ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος της ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωμένης Αριστεράς, Βόρειας Αριστεράς, η κυρία Σαΐμπη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε ο εξυγχρονισμός δεν θα πει ε, εργαζόμενοι μιας χρήσης. Ε, αυτό ονομάζεται επιστοφή στο μεσαίωνα. Παντού ε, στην Ευρώπη, στη Γερμανία, στην Αγγλία αλλά και στην παγκοσμίω, στη ΣΥΠΑ, στο Μεξικό η εκμετάλλευση γίνεται στους πιο ευάλωτους και μάλιστα καταδικάστηκαν ε, την περασμένη εβδομάδα κιόλα. Η δικαιοσύνη μάλιστα αναγνώρισε ότι υπό την προϋπόθεση, ε, υπό το πρόσχημα της ε, ευελιξίας ε, οι, κάποιες εταιρείες απασχολούσαν ποδηλάτες ως ανεξάρτητους επαγγελματίες και όχι ως υπαλλήλου. Ε, δηλαδή χωρίς καμία κάλυψη. Όλα αυτά μας αφορούν και σας αφορούν. Δεν μπορούμε να περιμένουμε πλέον. Τι περιμένουμε για να υποχρεώσουμε τις πλατφόρμες να αναγνωρίσουν ε, τους ε, ανθρώπους που κάνουν τις παραδόσεις ε, για αυτό που είναι, δηλαδή τους υπαλλήλου που πρέπει να έχουν την ίδια προστασία και την ίδια εκπροσώπηση ε, τη συλλογική όπως όλοι οι υπόλοιποι μισθωτοί. Σας ευχαριστώ και τώρα εξ ονόματος των μη εγγεγραμμένων μελών για ένα λεπτό ο κύριος Νικολάου Αλαβάνος. Παρακαλώ. Οι εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαρακτηρίζονται από έντονη ανησυχία για νέα ύφεση και κρίση. σε αυτό το περιβάλλον παρουσιάζεται σαν λύση μεταξύ άλλων την ψηφιοποίηση της οικονομίας. όμως στα πλαίσια της καπιταλιστικής οικονομίας αυτές οι καινοτόμες εφαρμογές γίνονται αντικείμενο έντονου ανταγωνισμού μεταξύ ευρωπαϊκών κινέζικων αμερικάνικων τεχνολογικών κολοσσών για το ποιο από αυτού θα προπορευτεί στην κούρσα κερδοφορία και με επιδοτήσει δισεκατομμυρίων ευρώ. αντί οι καινοτόμε εφαρμογέ να ανακουφίσουν τους εργαζομένους να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας θα ρίξουν στην ανεργία χιλιάδες εργαζόμενους σύμφωνα με τις δικές σας προβλέψεις θα τσακιστούν μισθοί θα διαλυθούν ωράρια συμβάσεις και ασφαλιστικά δικαιώματα. αυτή η αξεδιάλυτη αντίφαση είναι ίδιον του συστήματος της εκμετάλλευσης που με ζήλο υπερασπίζεστε και υπηρετούν η ευρωπαϊκή ένωση οι κυβερνήσεις της τόσο στην ελλάδα η νέα δημοκρατία σήμερα όσο και ο σύριζα προηγούμενα μόνο η εργατική εξουσία και η κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία αξιοποιώντα την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο είναι αυτή που θα λυτρώσει του λαού από τα βάσανα. αυτό είναι το μέλλον τη ανθρωπότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ένα λεπτό. Ε, κυρία Σχίδεντάλ, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια κοινωνική επιτυχία και η ενιαία αγορά είναι ο λόγος στον οποίο οφείλεται αυτό. Από τότε που η χώρα μου, η Σουηδία, μπήκε στην Ένωση πριν από 25 χρόνια, είδαμε μία ε, εξαιρετική άνοδο του ΑΕΠ μας, πράγμα το οποίο μας έχει δώσει την ευκαιρία να αυξήσουμε τις δαπάνες για την κοινωνική πρόνοια. Τα ημερομίσθια έχουν σχεδόν διπλασιαστεί και η κοινωνική πρόνοια είναι στο απόγειό τη. Το ίδιο επίσης σχήμα είναι ορατό στα νεότερα κράτη-μέλη. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να παίξει ρόλο όσον αφορά την κοινωνική πρόνοια εν μέρη μέσω νομοθετικών προτάσεων αλλά κυρίως μέσω της προώθησης μιας κοινωνίας, μιας μάλλον ε, αγοράς κοινωνικής πρόνοιας ε, και καθώ προκύπτουν νέε ευκαιρίε στον ψηφιακό κόσμο και μέσω τη ψηφοποίησης θα πρέπει να δούμε να, να αναδρομικά τι κάναμε και να διαρωτηθούμε πώ μπορούμε να το επαναλάβουμε. Θα πρέπει να αγωνιστούμε υπέρ κοινωνική πρόνοια ε, των ε, και ευημερία των συμπολιτών μας, όμως εάν λόγω κακής ρύθμισης ε, δεν τα καταφέρουμε, τότε δεν θα υπάρχουν ούτε νέες θέσεις απασχόλησης, ούτε κοινωνική πρόνοια για τους συμπολίτες μας. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ για ένα λεπτό. Ο κύριος Αγγιούς Σαλίμπα. Κύριε Πρόεδρε, ε, Επίτροπε, ναι, οι ψηφιακέ τεχνολογίε έχουν αλλάξει κάθε πτυχή τη ζωή μα, συμπεριλαμβανομένης των μοντέλων εργασίας και ε, ε, ε, επιχειρήν. Δεν υπάρχουν πραγματικά σύνορα, αλλά δεν υπάρχουν ούτε και ξεκάθαροι κανόνες. Οι ψηφιακές εταιρείες θέτουν νέους όρους, νέους κανόνες, ταράζουν τα νερά, διαφορετική όρια ασφάλειας και προστασίας των εργαζόμενων. Πρέπει να δώσουμε λοιπόν μια ισχυρή κοινωνική διάσταση και ένα ασφαλές επιγραμμικό το περιβάλλον για τους συμπολίτε μας. ότι δεν επιτρέπεται εκτός ε, του ίντερνετ δεν θα πρέπει να επιτρέπεται ούτε και στο ίντερνετ. Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται ε, να επιβαρυνθούν και να ζημιωθούν οι πολίτες. Θα πρέπει να προσέχουμε να αποφύγουμε την εκμετάλλευση των εργαζόμενων και επίσης ε, να υπάρχει και το δικαίωμα της αποσύνδεσης. Ε, όπως έχουν οι υπάλληλοι, έτσι θα πρέπει και να υπάρχει ένα μίνιμουμ χρόνου αποσύνδεσης ε, ημερησίως. Θα πρέπει λοιπόν να μελετήσει η Κομισιόν τους ψηφιακούς κινδύνους και τις συνέπειες της εργασίας αυτού του είδους για τους εργαζόμενους. Ευχαριστώ πολύ. Ανάμιση λεπτό η κυρία Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, κύριε Πρόεδρε, κύριε, ε, κύριε Επίτροπε, ε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου. Θα ήθελα να επιμείνω για τα εξή. Καταρχά, μία από τι πιο ορατέ συνέπειε τη ψηφοποίηση στον κοινωνικό τομέα και στον τομέα τη απασχόληση, και το έχουμε δει, είναι η εμφάνιση νέων ειδών εργασία μέσω των πλατφορμών. Αυτέ οι πλατφόρμε στην ουσία καλύπτουν πολύ διαφορετικέ πραγματικότητε, πράγμα που καθιστά πιο περίπλοκο το δικό μα έργο το νομοθετικό. Πρέπει να βρούμε την σωστή ισορροπία ανάμεσα στι και τι προοπτικέ απασχόληση και την προστασία αυτών των εργαζομένων αποφεύγοντα την ε, ε, επισφάλεια για αυτούς. Πρέπει λοιπόν να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην εργασία αλλά και στην κοινωνική κάλυψη σε σχέση με τις ασθένειες και τα ατυχήματα τα εργασιακά. Δεν έχω καμία αμφιβολία κύριε Επίτροπε ότι θα ασχοληθείτε με αυτό το ζήτημα. Πρέπει επίσης οι εργαζόμενοι να μπορούν να οργανωθούν συλλογικά για να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους. Ε, τέλος να μπορούν να ε, παρακολουθήσουν κατάρτιση επιμορφωτικά μαθήματα για να μπορούν να προοδεύσουν επαγγελματικά. Επίσης, κάτι που θέλω να τονίσω είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε πολύ άσχημη θέση όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες και ότι μόνο το 40% του εργατικού μας δυναμικού, μάλλον το 40% του εργατικού δυναμικού έχει από μηδενική πολύ ισχυρή γνώση των ψηφιακών δεξιοτήτων. Πρέπει αυτό να το διορθώσουμε ε, γιατί είναι ε, η 8η ε, ε, δεξιότητα κλειδί και θα πρέπει εκεί να επενδύσουμε όσον αφορά την επιμόρφωση. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό ο κύριος Λακαπέλ την εποχή ε, του 5G η περιφέρεια στη Γαλλία δεν έχει περάσει καν ακόμα στο ψηφιακό κόσμο. Έχουμε καθυστερήσει πολύ. Θα πρέπει να ξαναβρούμε μια Ευρώπη των εθνών και ο ψηφιακός κόσμος πρέπει να τεθεί στην υπηρεσία αυτών των εθνών. Η λογική της, ε, των έρθων συναλλαγμών γίνεται όλο και πιο ε, δημιουργεί όλο και με περισσότερες ανισότητες, γίνεται όλο και πιο άδικη. Ε, ανισότητες και μεταξύ φίλων και μεταξύ περιοχών και περιφερειών. Οι Μητροπόλεις αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα. Είμαστε εναντίον αυτού του άκρατου φιλελευθερισμού. Θέλουμε μια ευρωπαϊκή, δημοκρατική νέα Ευρώπη, η οποία θα είναι κοντά στους ανθρώπους, με, θα βασίζεται σε ε, κράτη-έθνη. Ευχαριστώ. Merci. Now for one minute. ευχαριστώ. Για ένα λεπτό, κυρία Ευχαριστώ. Η Κομισιόν μας υποσχέθηκε μια κοινωνική Ευρώπη. Και το έχει κάνει πολλές φορές για να γίνει αυτό θα πρέπει να δούμε τι αποτελέσματα έχει η ψηφιακή οικονομία. Το να βρει κανεί ε, προσιτή στέγη είναι σχεδόν αδύνατο σε πολλέ πόλει. Οι δήμαρχοι μεγάλων πόλεων όπω το Άμστερνταμ, η Πράγα, η Βαρκελόνη έχουν ε, πει ότι βασικός λόγος είναι το Airbnb και το Booking. Το Airbnb δεν φτιάχτηκε για να φτιάξουν οι επενδυτές παράνομα ξενοδοχεία, αλλά έχουμε φύγει ε, μακριά από την αρχική ιδέα του να νοικιάζει κανείς ένα κρεβάτι που του περισσεύει. Και αυτή τη στιγμή προστατεύονται τα δισεκατομμύρια των κερδών από το, παρά το δικαίωμα των ανθρώπων να έχουν προσιτή στέγη. Μιλάμε για κοινωνική Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε αυτό και όχι να ανοίξουμε την πίσω πόρτα έτσι ώστε οι μεγάλες ε, ψηφιακές εταιρείε να υπονομεύσουν την κοινωνική Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Για ένα λεπτό η κυρία Ντελαπίζα Καριών. Ευχαριστώ. Αναγνωρίζουμε την σημασία που έχουν οι ψηφιακές τεχνολογίες στη ζωή μας, ε, στο κοινωνικό μας και παραγωγικό μας μοντέλο πρέπει να πάρουμε σημαντικές προτάσεις για να προετοιμάσουμε το μετασχηματισμό. Η ψηφιοποίηση δεν επιτρέπεται να απανθρωπίσει τις κοινωνίες μας. Χρειαζόμαστε ένα καινούργιο εργασιακό μοντέλο και θα πρέπει ε, να αποφύγουμε η αυτοματοποίηση να οδηγήσει σε απώλεια θέσεων εργασίας. Η κατάρτιση, η επιμόρφωση των νέων θα πρέπει να γίνεται με ελαστικότητα και να του επιτρέπει να προσαρμόζονται στα νέα επαγγέλματα. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μια πραγματική και επαρκή προστασία των εργαζομένων εν ώψη αυτών των προκλήσεων. Ταυτόχρονα θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την ανταγωνιστικότητα τη επιχείρησή μα, την ανάπτυξή του και τι επενδύσει του. Είναι ευκαιρία να αναζωογονήσουμε τι περιοχέ τη υπαίθρου ε, μέσω τη πρόσβαση στην ψηφιοποίηση των κατοίκων του. Με αυτόν τον τρόπο θα αυξήσουμε την οικονομική, κοινωνική και ε, εδαφική συνοχή. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό, ο λόγος του κύριου Τζαρούσο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα πρέπει ε, κανείς να μην αποκλειστεί από τις ευκαιρίες της ε, ψηφιακής επανάστασης. Εκεί όπου υπάρχουν ανισότητες πρέπει να παρέμβουμε αμέσως για να μειωθούν αυτές, όχι να αυξηθούν. Το ίδιο ισχύει και για τους ε, επιχειρηματίες, όχι μόνο για τους πολίτες έχουν δημιουργηθεί ολιγοπόλια που σύμφωνα με την ευρωπαϊκή παράδοση πρέπει να ρυθμιστούν και να πληρώσουν τους φόρους που τους αναλογούν για να μην υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός ε, σε σχέση με την παραδοσιακή οικονομία. Τέλος, φάρμακα, γεωργία, πληροφορίες. Τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να είμαστε σε θέση να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες για να προστατεύουμε καλύτερα την υγεία, για να έχουμε καλύτερη γεωργία και προέλευση των προϊόντων μας και να καταπολεμούμε τις ψευδείς ειδήσει. Βεβαίως τα ψέματα διαδίδονται πολύ πιο γρήγορα στο διαδίκτυο, αλλά πολύ πιο εύκολα μπορούν να ξεσκεπαστούν κιόλα. Οπότε αυτό θα πρέπει να γίνεται με τρόπο γρήγορο, συνεχή και αποτελεσματικό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για ένα λεπτό κάζα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η τεχνολογία αλλάζει τις ζωές μας. Τον τρόπο που μελετούμε, τον τρόπο που εμπορευόμαστε, τον τρόπο που εργαζόμαστε. Έχουμε νέες ευκαιρίες αλλά ε, και νέες προκλήσεις. Ε, ε, Η οδηγία για την ισορροπία μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής ε, αναφέρεται σε όλα αυτά τα θέματα. Θα είναι θα είναι πιο εύκολο για τις γυναίκες να παραμένουν ε, στην αγορά εργασίας, αλλά και ε, θα είναι πιο εύκολο να μειωθούν οι διαφορές μεταξύ, στις αμοιβέ μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η Κομισιόν έχει μια στρατηγική την οποία καλωσορίζω, γιατί έχουμε, όπως είπαμε, νέες προκλήσεις. Το δικαίωμα στην αποσύνδεση θα πρέπει να είναι μέσα σε αυτό το νέο κανονισμό Χρειαζόμαστε νέες ασφαλιστικές δικλείδες και να εξασφαλίσουμε ότι αυτά τα δικαιώματα θα είναι προσιτά σε όλους. Ευχαριστώ πολύ και τώρα για ένα λεπτό η κυρία Τόγια. Ναι. Θα είναι σημαντικό να διατηρήσουμε στο νέα ψηφιακή ε, εποχή τις κοινωνικές και δημοκρατικές αρχές της Ευρώπης. Να δείξουμε δηλαδή ότι ο πολίτης είναι στο επίκεντρο όλων, αλλά πρέπει να το σκεφτούμε. Τα νέα μέσα δεν θα κάνουν αυτόματα αυτό το άλμα ποιότητα. Χρειάζεται σωστή πολιτική που να προσανατολίσει και να θέσει τους κατάλληλους κανόνες. Ε, δεν θα υπάρξει ψηφιακή δικαιοσύνη αν οι πολίτες και οι εργαζόμενοι δεν έχουν κατάρτιση και επιμόρφωση, όπως είπε και ο για τις νέες αυτές ε, ε, θέσεις απασχόλησης για τις οποίες πρέπει να, δικαιωθούμε, δικαιώματα, όπως ας για τους εργαζόμενους στις πλατφόρμες. Δεν θα υπάρξει κοινωνική και ψηφιακή δικαιοσύνη αν δεν θεσπίσουμε από τώρα τα μήνυμα νομικά μέσα για αυτούς τους ε, online εργαζόμενους που πρέπει, που, ε, πρέπει να ε, εργαστούν με αυτόν τον νέο τρόπο. Επίσης θα πρέπει τα κέρδη να, να φορολογούνται εκεί όπου δημιουργούνται και χρειάζεται γι' αυτό απόφαση του Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ένα λεπτό, Κάνιας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το 47% των θέσεων απασχόληση αυτή τη στιγμή ενδεχομένω θα χαθούν τα επόμενα 25 χρόνια και το 85% ε, του 2040 ακόμα δεν έχουν δημιουργηθεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η ψηφιακή οικονομία προσφέρει ευκαιρίες αλλά και έχει και, ενέχει και κινδύνους. Για παράδειγμα καινούρια χάσματα μεταξύ περιοχών, περιφερειών, φύλων κλπ. Τι μπορούμε να κάνουμε. Περισσότερη κοινωνική Ευρώπη, περισσότερη εκπαίδευση, επιμόρφωση, προστασία. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δούμε συνολικά το θέμα αυτό, σφαιρικά μέσω της Πράσινης ε, Συμφωνίας έχουμε αποφασίσει μια ε, αλλά, οικονομική αλλαγή της κοινωνίας μας, ε, της Ευρώπης. Γιατί όχι και μια ε, κοινωνική νέα συμφωνία, μια νέα κοινωνική συμφωνία, έτσι ώστε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν θα τα καταφέρουν χωρίς βοήθεια να ανέβουν στο τρένο του ψηφιακού μετασχηματισμού. Αυτό είναι ένας κίνδυνος τον οποίο θα πρέπει να αποφύγουμε για την κοινωνία μας. Ευχαριστώ. Gracias. Now for... Ευχαριστώ για ένα λεπτό ο λόγος του κύριο Ράιλ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι ιδιαίτερως για το ότι συζητάμε σήμερα για τις επιπτώσεις ψηφιοποίησης στην ε, κοινωνική Ευρώπη. Η ψηφιοποίηση βεβαίως ε, έχει ευκαιρίες αλλά και δυστυχώ μεγάλου κινδύνους. Πρέπει να δράσουμε. Να επενδύσουμε σε υποδομέ. Η Γερμανία έχει ένα από τα χειρότερα δίκτυα κινητή τηλεφωνίας στον κόσμο. Στη Γαλλία 13 εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν ίντερνετ ακόμα και πρέπει να μιλήσουμε και για την εκπαίδευση. Ο μισός πληθυσμός σχεδόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να χειριστεί τα ψηφιακά μέσα. Πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Αλλά με ανησυχούν ιδιαίτερα τα δικαιώματα των εργαζομένων στις πλατφόρμες. Δεν είναι δυνατόν να εργάζονται χωρίς δικαιώματα. Δεν τηρούνται ωράρια. Δεν υπάρχει καμία προστασία από απόλυση. Αυτά πρέπει να γίνουν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για ένα λεπτό κύριο Στανκανέλη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το ίντερνετ ε, από μία υποδομή των τηλεπικοινωνιών έχει γίνει ένα φαινόμενο με κοινωνικό ενδιαφέρον. Αλλάζουν οι, συνθήκη, οι συνήθειές μας, η καθημερινότητά μας και κάποιες πτυχές ε, οι οποίες ε, παρακολουθούνται συνεχώς, κάτι το οποίο μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις. Η απλότητα με την οποία μοιραζόμαστε το οποιοδήποτε περιεχόμενο είναι ένα πολύ ισχυρό όπλο στα χέρια οποιοδήποτε θέλει να εκμεταλλευτεί καταστάσεις οι οποίες δεν ρυθμίζονται. Γι' αυτό θα πρέπει να ασκούμε έναν συνεχή έλεγχο για τις ψηφιακές εφαρμογές έτσι ώστε αυτές να μην θέτουν σε κίνδυνο τις ατομικές ελευθερίες. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό η νομοθεσία να περιέχει σαφείς διατάξεις που θα εγγυώνται την ελευθερία του πολίτη, η οποία δεν πρέπει να είναι ένα απλό εμπόρευμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Και τώρα Κυρία Φράνσεν, για ένα λεπτό. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Το ψηφιακό χάσμα ε, διαχωρίζει όλο και περισσότερο αυτούς που έχουν ίντερνετ από αυτούς ε, που δεν μπορούν να εργαστούν. Και συνεχώς αυξάνονται οι learning, οι banking, η government και όλο και περισσότεροι άνθρωποι μένουν εκτός σκεφτόμαστε ε, αυτομάτως ε, ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ε, μεγάλη εκπαίδευση ή στερούνται οικονομικών μέσων. Και δικαίως, αλλά το χάσμα είναι κάτι ακόμη περισσότερο. Σήμερα ένας μηχανικός αυτοκινήτων πρέπει να ξέρει από υπολογιστές. 9 στις 10 νέες δουλειές χρειάζονται ψηφιακές δεξιότητες, αλλά 40% των Ευρωπαίων δεν έχουν επαρκή προσόντα. Γι' αυτό θα πρέπει να επενδύσουμε στις ψηφιακές δεξιότητες ε, των ανθρώπων και να προβλέψουμε εναλλακτικέ. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την ψηφιακή εκπαίδευση σε συνδυασμό με το Ταμείο της Παγκοσμιοποίησης έτσι ώστε όσοι χάσουν τη δουλειά τους να βρουν μια νέα. Ελπίζω λοιπόν η Κομισιόν να δώσει τις συμβουλές και να τις ακολουθήσει και το Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να λεπτό κύριος Βέλκιον. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Όταν μιλάμε για τις κοινωνικές πτυχές της ε, ψηφιοποίησης, ε, σκεφτόμαστε συχνά το εάν ε, το ίντερνετ είναι δημοκρατικός χώρος. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο η ελευθερία, αλλά και τα δικαιώματα των εργαζομένων η κοινωνική δικαιοσύνη στο διαδίκτυο για εμένα σημαίνει πρώτα απ' όλα ψηφιοποίηση ε, των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτό λοιπόν μπορούμε να κάνουμε. Να υπάρχει μια κυριαρχία του χρόνου, να υπάρχει περισσότερος χρόνος για την οικογένεια. Αυτό μπορεί να κάνει ψηφιοποίηση. Και πρέπει εδώ πέρα να υποχρεωθούν να δράσουν οι ψηφιακές πλατφόρμες. Δεν μπορεί να μην έχουν ευθύνη για τους εργαζόμενους τους. Και Πρέπει να δικτυωθούν και τα συνδικάτα. Και αυτό γίνεται πολύ καλύτερα μέσω ψηφιακών διάβλων. Η ψηφιακή Ευρώπη θα γίνει κοινωνική Ευρώπη όταν οι κοινωνικοί εταίροι ενισχυθούν και όχι μόνο τα κέρδη των μεγάλων εταιριών. Τώρα λοιπόν έχουμε την ευκαιρία σε όλες τις ε, επιτροπές ε, να δράσουμε από κοινού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Μελχιόρ για ένα λεπτό. Ε, Ο ψηφιακός κόσμος, το ίντερνετ, ε, έχει μετακινήσει τα εμπόδια, έχει εξαφανίσει τα εμπόδια στην εργασία ε, και έχει αμφισβητήσει πολλές εξουσίες εδώ και χρόνια. Δίνει καινούργιες ευκαιρίες, ενισχύει το άτομο, και δίνει περισσότερες δυνατότητες. Επίσης δίνει ευκαιρίες ε, εξειδίκευσης, ακόμα και στις περιοχές της υπαίθρου, να δημιουργηθούν καινούριες θέσεις ασίας, να αναζητηθούν καινούριες ευκαιρίες, εκεί που παλιότερα κάτι τέτοιο δεν θα ήταν δυνατό. Όμως απαιτεί υψηλή ποιότητα συνδέσεις ίντερνετ σε όλη την περιφέρεια. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να επεκταθούν οι υπηρεσίες αυτές και στις περιοχές της υπαίθρου, έτσι ώστε οι πολίτες μας να μπορούν να δημιουργήσουν τις δικές τους δουλειές. Θα πρέπει να δούμε και ποιες ευκαιρίες δημιουργούνται, όχι μόνο να βλέπουμε τις προκλήσεις. Έχουμε ένα κοινό κοινωνικό μέλλον στην Ευρώπη να φτιάξουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό ο Σφουρλας έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω και να καλωσορίσω όλους αυτούς τους νέους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω μας. Αυτή είναι το μέλλον της Ευρώπης, για αυτούς αγωνιζόμαστε το θέμα τη ψηφιακή μετάβαση είναι σημαντικό διότι μπορεί να ευκολύνει τι ζωέ όλων. ζητούμενο είναι μέσα από τι νέε ψηφιακέ τεχνολογίε να απλοποιήσουμε τι διαδικασίε προ όφελο του πολίτη και να διασφαλίσουμε ισότιμη πρόσβαση για όλου και ιδιαίτερα για τα άτομα που κινδυνεύουν από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. είναι ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσουμε ώστε να εντάξουμε καλύτερα και τα άτομα με αναπηρία στην αγορά εργασία να ανοίξουμε νέε θέσει εργασία είναι ευκαιρία που επίση δεν πρέπει να χάσουμε για να ενισχύσουμε την υγειονομική περίθαλψη. τα κράτη μέλη οφείλουν να προωθήσουν πολιτικέ που θα καταστήσουν τι δημόσιε υπηρεσίε πιο φιλικέ προ τον χρήστη αντιμετωπίζοντα δυναμικά τη γραφειοκρατία. κυρία πρόεδρε οι μισοί πολίτε μα εξακολουθούν να μην διαθέτουν βασικέ ψηφιακέ δεξιότητε. αυτό που οφείλουν τα κράτη μέλη είναι να προσαρμόσουν τα εκπαιδευτικά συστήματα στι νέε προκλήσει ώστε να μειωθεί το χάσμα που σήμερα υπάρχει στην ευρώπη ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Για ένα λεπτό λόγω στην κυρία Σάλντε Η ψηφιοποίηση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Κάποιος ο οποίος ε, έχει ένα ατύχημα στο σπίτι του μπορεί ε, να πάρει βοήθεια από το σπίτι του ε, ή κάποιος ε, μπορεί να πάει να μετακινηθεί χωρίς να οδηγήσει το αυτοκίνητό του στον προορισμό του. Ε, όμως έχουμε πάρα πολλούς εργαζόμενους οι οποίοι δεν έχουν ακόμα τα απαραίτητα προσόντα για να αγκαλιάσουν την ψηφιοποίηση. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα επηρεαστεί η προσωπική του ζωή, η ιδιωτικότητά τους επίσης. Θα πρέπει να καταλάβουμε πολύ καλύτερα πώς θα γίνονται οι επιλογές των καταναλωτών στο μέλλον μέσω του ίντερνετ και οπωσδήποτε χρειάζεται, χρειαζόμαστε μια ψηφιακή κοινωνία σύμφωνη με τις ανάγκες των ατόμων, όχι το αντίστροφο. Ευχαριστώ. Thank you very much. Now for one minute. Ευχαριστώ πολύ. Για ένα λεπτό λόγο στην κυρία Ντελκαστήγιο Βέρα. Η αρχική ερώτηση είναι τι είναι η κοινωνική Ευρώπη κοινωνική Ευρώπη είναι η Ευρώπη όπου κατά βάση όλοι έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσονται επαγγελματικά αλλά και να αναπτύσσουν την προσωπική του ζωή χωρίς να αποκλείεται κανένας. Αυτή είναι η ουσία της κοινωνικής Ευρώπης. Οι ψηφιακές τεχνολογίες προσφέρουν ακριβώς αυτό. Τη δυνατότητα ο καθένας και καθεμία από εμά να ε, πετύχει το στόχο του. Και τι χρειάζεται για να γίνει αυτό. Μία είναι η απάντηση, μία ιδέα η κατάρτιση, η εκπαίδευση, η ψηφιακή επιμόρφωση. Χρειάζεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, από την αρχή της ζωής των ανθρώπων, από την παιδική τους ηλικία, μέχρι τους ηλικιωμένους. Και χρειάζεται ένα πρόγραμμα δράσης για ψηφιακή κατάρτιση που να είναι πλήρες, σφαιρικό και σε αυτό θα πρέπει η Ευρώπη να ηγηθεί. Αυτό θα είναι το πιο σημαντικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Για ένα λεπτό λόγο στην κυρία Γκάλβες Η Ευρώπη θα πρέπει να προετοιμαστεί για την ψηφιακή επανάσταση χωρίς να αποκλειστεί κανένας, χωρίς να αποκλειστεί καμία περιοχή. Η ψηφιοποίηση θα πρέπει να ωφελήσει τους πάντες και να βοηθήσει έτσι ώστε να μειωθούν οι ανισότητες, να βελτιωθούν οι δημόσιες υπηρεσίες και να δημιουργηθούν νέες ποιοτικέ θέσει εργασία. Θα χαθούν πολλές θέσει εργασία, το ξέρουμε, αλλά θα δημιουργηθούν και πολλές καινούριε για παράδειγμα σχετικέ και συνδεδεμένε με, την τεχνητή νοημοσύνη. 58 εκατομμύρια θέσει εργασία αναμένεται να δημιουργηθούν εκεί πέρα. Όμω δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε τι γυναίκε. Μόνο το 22% των εργαζομένων σε αυτού του τομεί είναι γυναίκε. Υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ των δύο φύλων. Μόνο 22% των, ε, των εργαζομένων γυναίκε σε αυτού του τομεί. Χρειαζόμαστε μια σφαιρική εκπαίδευση και μια κουλτούρα, συνολική κουλτούρα που θα στηρίζει τα κατάλληλα προσόντα. Δεν μπορούμε επίσης να α, χάσουμε ούτε ένα ταλέντο. Τα ταλέντα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ε, υπάρχουν, αλλά δεν τους δίνονται επαρκείς ευκαιρίες και θα πρέπει να συνεργαστούμε έτσι ώστε αυτές οι ευκαιρίες να φτάσουν σε όλους και σε όλες, ιδίως στις γυναίκες. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό. Ο κύριος Μπέρεντσεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ψηφιοποίηση δίνει στην οικονομία μας πολλές ευκαιρίες μπορεί να ενισχύσει και την κοινωνία. Να βελτιώσει την υγεία, ασφαλείς μεταφορές. Όλα αυτά είναι δυνατά με την ψηφιοποίηση. Η αυξημένη ψηφιοποίηση της κοινωνίας όμως επιφέρει και τρεις κινδύνους. Καταρχάς, κανένας δεν πρέπει να μείνει ξεχασμένος, να μείνει πίσω. Όλοι θα πρέπει να ακολουθήσουν σε μια ψηφιακή κοινωνία. Και το περιβάλλον το σχολικό είναι πολύ σημαντικό εδώ. Δεύτερον, δεν θα πρέπει να αναπτύξουμε τεχνολογία σε κάποιες περιφέρειες και να ξεχάσουμε κάποιες άλλες. Πρώτα θα πρέπει να είναι οι λαοί και τρίτον η τεχνολογία θα πρέπει να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των λαών. Θα πρέπει να έχουμε ένα πλαίσιο για το τι είναι δυνατό και τι δεν είναι δυνατόν στην κοινωνία. Κανένας δεν θα πρέπει να ξεχαστεί. Δεν θα πρέπει να εξαρτώμαστε από άλλα μέρη του κόσμου και η τεχνολογία είναι υπέρ του λαού. Με αυτόν τον τρόπο θα προστατεύσουμε του πολίτε. Παράλληλα, θα υποφεληθούμε από τι τεράστιε ευκαιρίε που προσφέρει η τεχνολογία στην κοινωνία και την οικονομία μα. Ευχαριστώ για ένα λεπτό. Η κυρία Βίντ. Ευχαριστώ. Η τεχνολογική και ψηφιακή επανάσταση ε, αγγίζει όλα τα, τα τμήματα της ζωής μας. Το 2% του πληθυσμού εξασφαλίζουν το εισόδημά τους από την εργασία σε ψηφιακές πλατφόρμες και το νούμερο αυτό αυξάνεται καθώς περνάμε από το αναλογικό στο ψηφιακό επίπεδο. Πρέπει να έχουμε κατάλληλη νομοθεσία για τα, τους ελάχιστους μισθούς, τις συλλογικέ συμβάσεις, οι πλατφόρμες. Συχνά ξεχνάνε αυτές τις έννοιες. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε συνθήκες πληρωμής κατάλληλες για τους εργαζομένους. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι αρχές έχουν πρόσβαση σε, στους αλγόριθμους που χρησιμοποιούν αυτές οι πλατφόρμες. Αν θέλουμε να έχουμε μια ψηφιακή, αλλά και κοινωνική Ευρώπη παράλληλα. Ευχαριστώ. Α, ευχαριστώ. Για ένα λεπτό η κυρία Κάλερα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, Ακούσαμε εξαιρετικές ομιλίες ε, μέχρι τώρα. Ας ε, πιάσουμε την ουσία. Ως επιχειρηματίας της τεχνολογίας πληροφορίας και γυναίκα, πολλές φορές ε, μου έδωσαν καλοπροαίρετες συμβουλές, αλλά μετά από 15 χρόνια οι εργαζόμενοι μου και η εταιρεία μου δείχνουν κάθε μέρα ότι η ψηφιοποίηση δημιουργεί και εξασφαλίζει θέσεις εργασίας προφανώς επηρεάζονται και παραδοσιακές βιομηχανίες και κλάδοι. Στο Τυρόλο ε, ένα ξυλουργείο ε, τώρα επενδύει αντί να ανησυχεί για τους κινδύνους ε, και περνάει τη γραμμή παραγωγής από αναλογική σε ψηφιακή. Είχαμε κινδυνολογίες κατά το παρελθόν. παρόλα αυτά δεν απολύθηκε κανείς. Αντίθετα, αυξήθηκε το μερίδιο αγοράς και οι εργαζόμενοι. Αγαπητοί συνάδελφοι, έτσι βελτιώνεται η οικονομία και αυτό χρειαζόμαστε να προωθήσουμε, χρειάζεται να προωθήσουμε και εμείς οι πολιτικοί. Για ένα λεπτό, ο κύριος Γκαρσία Ντεμπλάνκο. Η ψηφιοποίηση, η εφαρμογή της τεχνητής νομοσύνης δηλαδή, προϋποθέτει μια, ε, σημαίνει μια τεράστια ευκαιρία. Πρακτικά θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα τεράστιο εξελεκτικό βήμα, το μεγαλύτερο μετά τη βιομηχανική επανάσταση. Βεβαίως ε, αυτό θα πρέπει να συνεπιφέρει αλλαγές και επίσης κάποιους φόβους, ανησυχίες που σχετίζονται με, ε, με, το, με την πιθανότητα απώλειας των θέσεων εργασίας και λοιπά, θέματα ασφάλειας. Ε, και υπάρχει και ένα άλλο θέμα, ο ψηφιακός αλφαβητισμός, δηλαδή η απόκτηση ψηφιακών ε, δεξιοτήτων, το οποίο συνεπάγεται μια ανθρωπιστική προσέγγιση στο θέμα, ούτω ώστε να εφαρμοστούν ζητήματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη και οι πολίτες αποκτήσουν επίγνωση των ε, κινδύνων και των αξιών που διακυβεύονται εδώ τους ώστε να μπορέσουν να λάβουν καλύτερες αποφάσεις στο πλαίσιο μιας ε, κοινωνίας η οποία είναι όλο και πιο ολοκληρωμένη. Γι' αυτό ζητώ από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να καταβάλουν ε, κάθε δυνατή προσπάθεια ούτω ώστε να μπορέσουν ε, όλα αυτά να τα μετασχηματίσουν σε κάτι εφικτό και προσιτό από όλους. Ευχαριστούμε.